και το Συμβούλιο, το ώστε όλοι να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε καλή δουλειά. Ξανά ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, εισηγητή. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση. Ε, αύριο στις 12 θα έχουμε την ψηφοφορία. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο θέμα της μερίσης διάταξης. Πρόκειται για την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά ε, για με την αποδοχή της προσχώρησης 8 τρίτων χωρών στη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για αστικά θέματα της διεθνούς απογωγής παιδιών. Ε, δίνω ε, τον λόγο στην εισηγήτρια, κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Είμαι ε, τώρα εκπρόσωπος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για τον κύριο Στογιάννοφ. Ε, τα αστικά θέματα στην απαγωγή των παιδιών ε, ε, υπάρχει η σύμβαση της Χάγης η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία έτσι ώστε ε, τα ε, παιδιά να μπορούν να επανέρχονται στο τελευταίο τους χρόνο διαμονής. Η Κομισιόν ε, μπόρεσε να ακολουθήσει το σωστό δρόμο στην προσφόρηση του Μαρόκο, της Ρωσίας, της Ανδόρας, της Σιγκαπούρης, της Αρμενίας και άλλων χωρών να μπουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοιπόν, έχουμε την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις εξωτερικές υποθέσεις. Εξωτερική αρμοδιότητα. Έχουμε την κανονισμό Βρυξέλλες 1 για την ε, αμοιβαία αναγνώριση της διεθνούς δικαιοδοσίας και της εκτέλεσης της εκτέλεσης αποφάσεων, ε, το οποίο είναι ξεκάθαρο προς τις αρμοδιότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλάμε για διεθνείς απαγωγές, Έχουμε την ε, εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αποκλειστική αυτή αρμοδιότητα. Το Συμβούλιο είχε ε, όμως μπλοκάρει αυτό το θέμα εδώ και καιρό και πρέπει να σταματήσει αυτό και πρέπει να διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών, πάντοτε αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Ε, όλο και περισσότερο μόνο το κοινοβούλιο ασχολείται με τα θέματα των ε, ε, πολιτών. Εμείς δεν βλέπουμε λόγο γιατί να μην προσχωρήσουν οι χώρες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν θέτω το ερώτημα στην Κομισιόν. Γιατί το Συμβούλιο πλοκάρει μια τόσο πολύ σημαντική απόφαση. Είναι πολύ σημαντική η προσχώρηση των τριτών χωρών το πόσο σημαντική είναι η προχώρηση το δείχνουν ξεκάθαρα τραγικέ υποθέσεις που βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απαγωγές παιδιών ε, ε, σε χώρες όπως η Αυστρία από όπου προέρχομαι. Ε, έχουμε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τρίτες χώρες και αφορούν οικογενειακές τραγωδίες. Ο Όλιβερ Χάρτλιν βρίσκεται με τον πατέρα του στην Δανία. Η μητέρα και οι παππούδες ε, λυπούνται γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει στην Αυστρία. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές απόψεις σχετικά ε, με την ε, απαγωγή εντό εισαγωγικών αυτού του παιδιού ε, μεταξύ της Δανίας και της Αυστρίας. Από τη μία δεν θεωρείται απαγωγή η συμπεριφορά του παιδιού και από την άλλη θεωρείται. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά ε, χώρες όπως η Ρωσία και το Μαρόκο, έχουμε πάρα πολλούς Ευρωπαίους πολίτες ε, που έχουν οικογενειακές σχέσεις με αυτά τα κράτη. Έχουμε παρόμοιες περιπτώσεις, ε, λοιπόν, με αυτή του Όλιβερ που δείχνει ακριβώς πόσο σημαντική για την ευημερία του παιδιού είναι η προσχώρηση των κρατών αυτών στη Συμφωνία. Ευχαριστούμε την συνάδελφο για τη σύνοψη αυτής της θέσης. Ε, η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που έφυξε το σημαντικότατο αυτό ζήτημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η επαγωγή των παιδιών από τους γονείς είναι μια τραγωδία. Πολύ συχνά έχει μακροπρόθεσμες ουσιαστικές συνέπειες για το παιδί. Και η πρόληψη αυτής της αρπαγής των παιδιών θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την πρόθεση των δικαιωμάτων των παιδιών. Και σε διεθνείς περιπτώσεις πολυμερείς κανόνες είναι βασικοί για να εξασφαλίσουν την προστασία των παιδιών. Από το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρες μέλος της διασκέψεως της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και σε αυτό το πλαίσιο η Ένωση υποστηρίζει την σύμβαση της Χάγης του 1980 για τις πολιτικές ε, για τις αστικές τυχές της απαγής παιδιών και ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή τη σύμβαση. 87 συμβαλόμενα μέρη είναι σήμερα στη Σύμβαση της Χάγης, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Σύμβαση θεσπίζει ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ των συμβαλωμένων μερών για την αποκατάσταση του status quo ante ε, του παιδιού που έχει ε, αποτελέσει δικείμενο αρπαγή. Αλλά για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα πρέπει να υπάρξει ρητή δήλωση αποδοχή. Και γι' αυτό πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη μέτρων για την αποδοχή από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω οκτώ νέων συμβαλωμένων μερών στη σύμβαση. Συμπαραβαμένων βασικών εταίρων όπω είναι η Ρωσία και το Μαρόκο. Η έγκριση τέτοιων προτάσεων θα εξασφάλιζε το ότι όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό της Χάγης με όλα τα συμβαλόμενα μέρη της συμβάσεως για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις απαγωγής παιδιών και αυτό θα ήταν προς το καλύτερο συμφέρον των παιδιών και θα σεβόταν και την αρχή της ενότητας όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά, λυπούμε. Λυπούμε που αυτό το πακέτο έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Ένα χρόνο έχει κολλήσει περίπου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η προσχώρηση της Σιγκαπούρης έγινε δεκτή από 10 κράτη-μέλη, του Μαρόκου από 14, των Σεϊχελών από 18 κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει επίσης ότι αφού επί σειρά ετών υπερασπιστήκαμε την προσχώρηση της Ρωσίας και αφού πείσαμε τη Ρωσία να προσχωρήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της τώρα δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την προσχώρηση. Και οι ρωσικές αρχές βεβαίως μας το θέτουν στις τακτικές συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Λυπούμε βαθύτατα. Λυπούμε διότι παρά τις δηλώσεις προθέσεων από πλευράς κρατών μελών, τα κράτη-μέλη στο σύνολό τους απέτυχαν μέχρι τώρα να δείξουν την κατάλληλη ευαισθησία και την πολιτική προθυμία που απαιτείται ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί η κατακαιρματισμένη αντιμετώπιση που υπάρχει όσον αφορά ε, τις την απαγωγή των παιδιών σε διεθνές επίπεδο και φοβούμε ότι ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί όσον αφορά την διοργανική αυτή διαφορά περί αρμοδιοτήτων που έχει πολύ ανεπιθύμητες συνέπειες και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Λίχτενμπέργκερ διότι υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εν γέννη που επεξεργάστηκε το θέμα. Έχουμε όλοι μας αισθανόμαστε την κοινή ανάγκη να προστατεύσουμε τα παιδιά, να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο και να μειώσουμε και τα και τα προβλήματα που περνούν οι οικογένειες λόγω ελλείψους ασφάλειας δικαίου και ελλείψεως ενωπημένων νομικών διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέμα. Και πραγματικά λυπάμαι γιατί έχουμε κολλήσει και πολεμάμε για διαδικασίες αντί να πολεμάμε για το καλό των παιδιών. Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο για τα ξεκάθαρα λόγια της. Το, το λόγο έχει η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια και την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ. Ξεκινώντας από ένα γεγονός. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σταδιακά η κυκλοφορία των προσώπων αυξάνονται συνεπώς και οι γάμοι και οι ενώσεις και από την άλλη πλευρά αυξάνονται και τα διαζύγια και οι χωρισμοί ε, ζευγαριών από διαφορετικέ χώρε. Περίπου 300.000 ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων παντρεύονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Το μισό περίπου από τους γάμους καταλήγει σε διαζύγιο ή χωρισμό. Αυτό, αυτή η διαμάχη και ο χωρισμός πολύ συχνά οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες ε, για τα παιδιά. Που τα διεκδικούν τα παιδιά όχι μόνο οι δύο γονείς, αλλά και δύο διαφορετικές χώρες και δύο διαφορετικά νομικά συστήματα. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό, μεταξύ άλλων, είναι σημαντική σύμβαση της Χάγης που υπεγράφει από 87 κράτη και από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολυμερείς συμφωνίες για την προστασία των ανηλίκων καθορίζει βασικούς κανόνες και θεσπίζει σαφή κριτήρια κυρίως όταν ο ανήλικος κινδυνεύει να μεταφερθεί και να, σε άλλη χώρα και να μην επιστρέψει στη χώρα συνήθως διαμονής. Προστατεύονται τα παιδιά τα ανήλικα από αυτές τις διαφορές όπου μπορούν τα παιδιά να γίνουν πραγματικά θύματα αυτών των εντόνων διαφορών. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό και απεχθές ότι η σχετική διαδικασία για την προσχώρηση 8 κρατών στη Σύμβαση της Χάγης έχει μπλοκαριστεί από το Συμβούλιο. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, για να δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε νέες απαγωγές παιδιών που αφορούν τη Ρωσία που είναι από μία από τις χώρες που ε, έχει κάνει διακήρυξη αποδοχής. Μία προσχώρηση της Ρωσίας είναι κάτι περιμέναμα από καιρό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μου, η οικογένεια είναι βασική ε, αξία για την κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα πρέπει να τη βοηθήσουμε, να την προστατεύσουμε. Τα θεσμικά όργανα προστατεύσουν την οικογένεια, κυρίως στιγμές που περνά κρίση η οικογένεια. Με βασικό σκοπό να προστατεύσουμε τα ανώτερα συμφέροντα των ανηλίκων, το να μπλοκάρεται μια διαδικασία που θα έπρεπε να ζητά επιτάξει των διαδικασιών, όχι μόνο αρνείται την προώθηση αυτών των στόχων, δηλαδή να έχουμε πιο εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, αλλά πάνω απ' όλα στην πραγματικότητα αρνούμεθα την προστασία των συμφερόντων των ανηλίκων. Εν κατακλείδη και σαν διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περιπτώσεις διεθνών απαγωγών, γνωρίζω ότι πολύ μεγάλος αριθμός περιπτώσεων προκύπτει από την αβεβαιότητα για το δίκαιο που ισχύει, από σύγκρουση δικαιοδοσιών, από ανεπάρκεια γνώσεων και γνώση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ζευγαριών που είναι από διαφορετικές χώρες οι δύο Ευχαριστώ συνάδελφε. Ε, για λόγους ε, που δεν γνωρίζω, η εκπρόσωπος των φιλολευθέρων δεν μπορεί να είναι εδώ ε, για να μιλήσει, οπότε δίνω το λόγο στην κυρία Λίχτενμπεργκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μένα αυτό το θέμα δείχνει την παρελκυστική πολιτική του Συμβουλίου. Ε, ε, θεωρώ ότι πρέπει να την καταδικάσουμε. Η απαγωγή των παιδιών από μόνη είναι ένα τραυματικό γεγονός, ένα βίωμα για το παιδί τουλάχιστον, πόσο μάλλον για, το, για τους γονείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουν ότι τουλάχιστον οι νομικές δυνατότητες ε, ε, θα βελτιωθούν έτσι ώστε το, παιδί να μπορέσει όσο το δυνατό γρηγορότερα να γυρίσει εκεί που αισθάνεται καλύτερα, εκεί που έχει συνηθίσει. Η σύνθεση της Χάγης είναι ένας τέτοιος μηχανισμός ε, που σε τέτοιες περιπτώσεις περι... προασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών και δίνει ε, βοήθεια σε διμερείς ε, περιπτώσεις απογωγής παιδιών. Έχουμε λοιπόν ε, δύο τώρα εταίρους την ουρά, τη Ρωσία και το Μαρόκο, που όλο και περισσότερες περιπτώσεις δύσκολες αντιμετωπίζονται και θα μπορούσαμε αυτό το πρόβλημα αύριο και μόλις να το διευκολύνουμε για τους εμπλεκόμενους εάν το Συμβούλιο ε, πραγματικά άφηνε και είμαι ξεκάθαρη σε αυτό στην άκρη αυτό το παιχνίδι που παίζει, ε, το παιχνίδι δυνάμεων. Το Συμβούλιο δεν θέλει την ε, συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα. Δεν συνεννοείται σε θέματα τόσο συγκεκριμένα και γι' αυτό οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύμβαση της Χάγης με αυτά τα κράτη τα τρίτα κράτη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πόσα παιδιά, πόσοι γονείς ήδη έχουν ε, υποστεί βλάβη λόγω αυτής της παρελκυστικής πολιτικής του Συμβουλίου. Κάνω έκκληση λοιπόν στο Συμβούλιο να μπλοκάρει κάτι άλλο. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Αφήστε μας λοιπόν ε, να προχωρήσουμε κανονικά με την συμμετοχή του Κοινοβουλίου όπως θα πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την συνάδελφο. Η κυρία ε, Ματίνα Άντερσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Οι τρομακτικές εικόνες από τη Γάζα μας υπενθυμίζουν δυστυχώς ότι είναι τα ευπαθέστερα άτομα τα παιδιά ακόμη και όταν βρίσκονται στο κέντρο της διεθνούς προστασίας. Θα πρέπει να αποκτήσουν πολύ πιο κεντρικό ρόλο στη, σε όλα τα επίπεδα κατά την κατάρτιση νέων νομοθετημάτων ε, τα παιδιά διότι δεν ακούγονται οι φωνές τους από τόσες πολλές πλευρές. Οι πολιτικές που ακολουθούνται από τις κυβερνήσεις και που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν σε αναρρύθμιτες σε περιπτώσεις αμελίας εις βάρος των παιδιών. Αυτό κατεδείχθη στη διάσκεψη την περασμένη Παρασκευή στο Belfast για τα παιδιά. Στι 10 Νοεμβρίου η Ιρλανδία ψήφισε για τροποποίηση συντάγματό τη, ώστε να διαφυλάξει τα δικαιώματα των παιδιών. Χρειάζονται όμω και πόροι από πλευρά τη κυβέρνηση για το Κέντρο προστασία και υποδοχή των Παιδιών και των Οικογενειών του. αλλά τουλάχιστον κάναμε ένα βήμα σε σχέση με τι διεθνεί μετακίνησει και τι νέε διεθνεί εξελίξει. Θα έλεγα ότι παρατηρείται ένα ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό απαγωγών παιδιών και γι' αυτό η Σύμβαση της Χάγης σε σχέση με τις διεθνείς απαγωγές σε παιδιών συνιστά πολύ σημαντικό κομμάτι της διεθνούς αρχιτεκτονικής για την προστασία των παιδιών καθότι προβλέπει την ταχεία επιστροφή των ε, απαχθέντων παιδιών στις χώρες ε, προέλευσης τους. Όμως υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με τον ε, ρυθμό, δηλαδή χρειάζονται χρόνια για να λυθούν υποθέσεις και άλλες παραμένουν άλυτες. Λόγω εξαιτία του Συμβουλίου παρεμποδίζεται η πρόσβαση τρίτων χωρών στη Σύμβαση και πρόκειται για σκάνδαλο. Πρέπει να αποτραπεί αυτή η κατάσταση, διότι χωρί απολύτω κανένα λόγο εκθέτουν τα παιδιά σε αυτόν τον κίνδυνο ε, και δεν παρεμποδίζουν τι διεθνεί απαγωγέ παιδιών ε, εξαιτία αυτή τη στάση του. Σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο, ο κύριο Τσίφκα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι είναι όντως ιδιάζουσα. Συζητούμε για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα και είναι πάρα πολύ θετικό που θέλουμε να εγκριθούν οι νέοι μηχανισμοί και μας παρεμποδίζουν οι διαθεσμικές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πρόκειται για σκάνδαλο η σημερινή μας συζήτηση είναι ουσιαστικά μια έκκληση προς το Συμβούλιο για να σοβαρευτεί επιτέλους και να χειριστεί με ε, τη δέουσα σοβαρότητα την τραγική κατάσταση τόσων ε, γονέων και παιδιών. Αν πίστευα στις θεωρίες συνωμοσία θα έλεγα ότι ε, δημιουργεί εκ του πρόβλημα στο Κοινοβούλιο του Συμβούλιο για αυτό το πράγμα. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρη όταν απεφάνθη Ανέφερε στη γνωμοδότησή της ότι υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα διεθνούς απόγεισος. Εκ τούτου το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο από κοινού θα πρέπει να εγκρίνουν σχετικές αποφάσεις. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να πείσουμε τρίτες χώρες για να προσχωρήσουν σύμβαση της Χάγης. Πρόκειται για μια αργή διαδικασία, ούτως ή άλλως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και απευθύνω θερμή έκκληση προς όλους όσους έχουν κάποια επιρροή. Ας μην παρακολύουμε την έγκριση ε, τόσο πρόσφορων λύσεων. Τα συμβαλόμενα μέρη που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε αυτή τη διεθνή συμφωνία δεν πρέπει να παρεμποδιστούν. Ας αφήσουμε τις τρίτες χώρες να επικυρώσουν τη σύμβαση γιατί έτσι ενισχύεται η ένομη τάξη ε, για ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα όπως οι διεθνείς απαγωγές. Ελπίζω μάλλον ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία γιατί θα γελιοποιηθούμε αλλιώς Γι' αυτό το λόγο, ξαναλέω, το Κοινοβούλιο πρέπει να απευθύνει έκκληση προς το Συμβούλιο για να αρχίσει να επεξεργάζεται μια ικανοποιητική λύση. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε δύο ε, βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Φασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς η παράνομη απαγωγή παιδιών και κράτηση των παιδιών δεν είναι με κάτι απομονωμένα. Όταν χωρίζουν οι γονείς υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την επιμέλεια των παιδιών και, και την κυδεμονία των παιδιών. Και πολύ συχνά αποφασίζουν να, φύγουν, να φύγει ένα γονέα γονέας από μια χώρα με το παιδί χωρί τη σύμφωνη γνώμη του άλλου. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Πριν την σύμβαση αυτή, πολύ συχνά τα παιδιά έπρεπε να επιστραφούν λόγω δικαστικών διαφορών μεταξύ χωρών. Υποχρονόταν να ζουν τα παιδιά σε ξένο περιβάλλον και αυτό οδηγεί σε κοινωνικές δυσλειτουργίες ε, και γλωσσικές δυσλειτουργίες, πολύ σοβαρές μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν την προσχώρηση των κρατών αυτών στα, στη σύμβαση. Ε, Κυρία Επίτροπη, ξέρετε πόσες ε, περιπτώσεις επηρεάζονται από αυτή την καθυστέρηση για την έγκριση των νέων προσχωρήσεων και τι μέτρα σκοπεύει να λάβει η Κομισιόν για να λυθεί το πρόβλημα. Ζητώ συγγνώμη που ήρθα τόσο αργά σε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Αντιπρόεδρε Ρέντινγκ, Είμαστε σε πάρα πολύ καλή επαφή για ένα θέμα, για τον Όλιβερ Βάιχαλ, ένας Αυστριακός πολίτης ο οποίος απήχθηκε, βρέθηκε στη Δανία. Η απαγωγή παιδιών, είτε πρόκειται για εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το χειρότερο αδίκημα και αν ε, ε, ε, έχουμε παρακολήσεις και δυσκολεύουμε την κατάσταση για τέτοια παιδιά πραγματικά χρειάζεται άμεση δράση σε διεθνές επίπεδο. Είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς μπορούμε να, να λειτουργήσουμε διεθνώς αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που ζητά το λόγο ε, στη διαδικασία Catch the Eye. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Επίτροπο Ρέντινγκ για τις τελικές παρατηρήσεις. Πρόεδρε, δεν περίμενα λιγότερα από το Κοινοβούλιο και από αυτά που εξέφρασε σαφέστατα το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, έχω συγκλονιστεί τα μάλα. Θα μπορούσε να επιλεγεί οδήποτε, ε, θέμα για μάχη μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων, αλλά όχι τα παιδιά. Και ακόμα και αν η ζωή ενός παιδιού επηρεαστεί από αυτή τη διαμάχη τη οργανική, αυτό είναι μια ζωή παραπάνω που κινδυνεύει. Η ζωή των παιδιών διακυβεύεται εδώ και θα πρέπει να σταματήσουμε τα παιχνίδια. Αυτό είναι το μήνυμα που έχω να στείλω στα κράτη-μέλη και ελπίζω να εισακουστεί το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που με βοηθάτε να πολεμήσω σε αυτή τη μάχη που δίνω. Ευχαριστώ. Ε, με αυτήν ε, την τελική θέση κλείνει η συζήτηση. Αύριο στις 12 η ώρα έχουμε την ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ε, την έκθεση